αλλά ιδιαίτερα να επαγρυπνούμε. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ειδήσει καν για την ε, υγεία του Προέδρου Ετζαλάν. Πρέπει να επαγρυπνούμε πάντα για να βοηθούμε τον κουρδικό λαό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Φορέντσα. Έχουμε λάβει ορισμένα αιτήματα για τροποποίηση, ε, αλλαγέ στα ονόματα και τους διορισμούς της Επιτροπές και τις Αντιπροσωπείες. Έχετε τα σχετικά στοιχεία στα έγγραφα της τρέχουσας συνεδρίασης. Αν δεν εκφραστούν ενστάσεις μέχρι την έγκριση των πρακτικών θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται και οι διορισμοί. Και τώρα προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε τον προπολογισμό.